Colleagues, uh, Συνάδελφοι, αρχίζουμε με τις ανακοινώσεις. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να αρχίσουμε τις ψηφοφορίες. Λοιπόν, αρχίζουμε με το γλωσσικό. Τους γλωσσικούς συνδυασμούς θα έχετε διερμηνία σε όλες τις γλώσσες εκτός από τα κρατικά και τα γκέλικ. Τώρα, έγκριση των συστάσεων των συντονιστών βάσει του άρθρου 205, ορισμός εισηγητών. Η κυρία Μπακασαρντουντού Αρουίθ από το ΑΛΔΕ είναι η συγγήτρια γνωμοδότηση όσον αφορά την πρόταση οδηγίας για την προστασία των προσώπων και τις παρεμβάσεις του νοσιακού δικαίου. Λάνερς ορίστηκε συγγητής για τροποποιημένη πρόταση όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύνορα και λοιπά. Μέλο όσον αφορά τον κανονισμό που ορίζει πλαίσιο για τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των Ευρωπαϊκών Στημάτων Πληροφοριών, Αστυνομία, Δικαστική Συνεργασία, Σύλλο και Μετανάστευση. Η Επιτροπή μας συμφωνεί. Ναι. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία σε λίγο. Καθίστε και ετοιμαστείτε παρακαλώ. Όλες οι ψηφοφορίες είναι ηλεκτρονικά. Αν δεν έχετε την ε, κάρτα σας, να το πείτε τώρα παρακαλώ. Εντάξει, έχετε όλοι τις κάρτες σας για να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Θα αρχίσουμε λοιπόν σε λίγο, εφόσον είμαστε όλοι έτοιμοι.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 σχεδίου έκθεσης ε, για το οποίο συγγήτρια είναι η κυρία Σαρτζεντίνη. Θέλετε να πείτε κάτι κυρία Σαρτζεντίνη? Όχι, ωραία. Αρχίζουμε λοιπόν με την ψηφοφορία. Έχω μία ανακοίνωση. Η κυρία Γκυγιόμ δεν έχει συνυπογράψει την τροπολογία 253, οπότε θέλει να αφαιρεθεί το όνομά τη από την τροπολογία αυτή 253. Με αυτήν την ε, τροποποίηση λοιπόν αρχίζουμε την ψηφοφορία. Συμβιβαστική τροπολογία 7. Ψηφίστε παρακαλώ. Ηλεκτρονικά. Ψηφίστε, γιατί βλέπω ότι ακόμα έρχονται διάφοροι και κάθονται. Καθίστε λοιπόν, ψηφίστε. Και συγχρόνως όσο παραμένει ανοιχτή ψηφοφορία να σας πω ότι έχουμε έναν παραπάνω από το ΕΛΚ που ψηφίζει. Οπότε πρέπει να αφαιρεθεί μια κάρτα. Τώρα είναι εντάξει. Ωραία. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 8. Ψηφίστε. Πέρας. Οι σοσιαλιστέ τώρα έχουν ένα παραπάνω που ψηφίζει. Ας αφαιρέσει κάποιο την κάρτα του παρακαλώ. Να αποσυρθεί μία κάρτα παρακαλώ. Ωραία. Πέρα τη ψηφοφορία εγκρίθηκε. Συμβαστική 9. Ψηφίστε. Συμβαστική 9. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά πέρα τη ψηφοφορία. Α, όχι, το ΕΛΚΑ έχει ένα παραπάνω. Εντάξει, ξέρω ότι όλοι είσαστε πολύ πρόθυμοι να ψηφίσετε σήμερα, αλλά το ΕΛΚ πρέπει να αφαιρέσει μια κάρτα, παρακαλώ. Ωραία, έγινε. Τώρα, πέρα τη ψηφοφορία. Και εγκρίθηκε. Συμβαστική 10. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 11. Ψηφίστε. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 12. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 13. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 38 τώρα. Δεύτερο τμήμα. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 14. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 15. Ψηφίστε. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 16. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 17. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 18. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. 19. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 20. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 25. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 27. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 28. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε. 29. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 90 τώρα. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 94 τώρα. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Απορρίφθηκε. Συμβιβαστική 30 τώρα. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 110 τώρα. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 111. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Απορρίφθηκε. Συμβιβαστική 35 τώρα. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 123. Ψηφίστε. Πέρασε. Απορρίφθηκε. Συμβιβαστική 37, λέει ο πρόεδρος. συγγνώμη, διορθώνει 36. Συμβαστική 36. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 37 τώρα, ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 38. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 39. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 41. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 42. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 43. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 154 τώρα. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας και απορρίφθηκε. Συμβιβαστική 44 με προφορική τροποποίηση. Ψηφίστε. Πέρα τη ψηφοφορία και εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 45. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Συμβαστική 46. Ψηφίστε. Μια στιγμή. Θέλετε να επαναλάβουμε την ψηφοφορία για τη συμβαστική 45. Γιατί έγιναν λάθη. Λοιπόν, κάποιοι ζητούν επαναληφθεί ψηφοφορία για την τροπολογία 45. Μια στιγμή, ηρεμήστε. Έχετε διαδικαστικό. Ωραία. Παρακαλώ και σύντομα. Πρόεδρε, το πρόβλημα είναι ότι η ψηφοφορία δεν ανακοινώθηκε σωστά μετά από την προηγούμενη. Ωραία, λέει ο πρόεδρο. Εντάξει, λοιπόν, ψηφίζουμε τη συμβαστική 45. Μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά. Κύριε Γιούρεκ. Ο κύριος Γιούρεκ. Πρόεδρε, βάσει ποιου επιχειρήματος θα επαναλάβουμε την ψηφοφορία, μπορείτε να μου πείτε. Γιατί θα την επαναλάβουμε αυτή την ψηφοφορία. Γιατί στην Ολομέλεια πολλές φορές ζητάμε να επαναληφθεί κάποια ψηφοφορία. Ακόμα και οι μεγάλες πολιτικές ομάδες το ζητούν, αλλά κάθε φορά απορρίπτονται τα αιτήματα αυτά. Όχι επειδή σε κάποιον δεν αρέσει το αποτέλεσμα, επαναλαμβάνουμε την ψηφοφορία. Πρόεδρος, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό αλλά δύο τουλάχιστον πολιτικές ομάδες είπαν ότι δεν είχαν καταλάβει ακριβώ τι ψηφίζανε. Οπότε γι' αυτό θα ξαναψηφίσουμε για τη συμβαστική 45. Έπειτα στη μέση της ψηφοφορίας ζητάτε διαδικαστικό, καλύτερα πρώτα να γίνεται η ψηφοφορία και μετά το διαδικαστικό. Λοιπόν, συμβαστική 45, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ, ηλεκτρονικά. Ο κύριος Γιούρεκ δεν βλέπω που αναφέρεται αυτή η αβεβαιότητα που λέτε. Συμβαστική 45, λέει ο πρόεδρος. Ψηφίστε. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 46. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 169 τώρα. Πρώτο τμήμα. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Συμβιβαστική 48. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 48α. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 49. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 178. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίστε παρακαλώ. 178 δεύτερο τμήμα. Ψηφίστε πέρασε τη Απορρίφθηκε. Τροπολογία 202, πρώτο τμήμα. Ψηφίστε παρακαλώ. «202 πρώτο τμήμα». Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Τρίτο τμήμα τώρα της 202. Τρίτο τμήμα, ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Απορρίφθηκε. Συμβαστική 50. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 186. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 188. Με μια προσθήκη. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Απορρίφθηκε. Συμβιβαστική 51 τώρα. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 52. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 53. Ψηφίστε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 54. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της υποφορίας Εγκρίθηκε. Τροπολογία 208. Ψηφίσουμε μόνο την προστίκη. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της υποφορίας απορρίφθηκε. Τροπολογία 210. Ψηφίστε. Πέρας. Απορρίφθηκε. Συμβαστική 55. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 212. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Απορρίφθηκε. Συμβαστική 56. Ψηφίστε. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 216. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκε. Συμβαστική 57. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 220. Μόνο την προστική ψηφίζουμε. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκε. Συμβαστική, 58. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 59. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 233. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκε. Συμβιβαστική 60 τώρα. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 61. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 244. Μόνο την προσθήκη ψηφίζουμε. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκε. Συμβαστική 62. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 247 τώρα. Ψηφίζουμε την προσθήκη μόνο. Ε. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 257. Μόνο την προσθήκη. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 164. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίστε. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 250. Ψηφίστε. Πέρας. Εγκρίθηκε. 253. Ψηφίστε. Πέρας. Απορρίφθηκε. Συμβαστική 1 από τις αιτιολογικές αναφορές. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα. Εγκρίθηκε. 2. Ψηφίστε. Πέρασε. Εγκρίθηκε συμβαστική 3. Ψηφίστε. Πέρας. Και εγκρίθηκε 4. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 6. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 21. Την προσθήκη. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Απορρίφθηκε. Πάμε στην τελική ψηφοφορία με ονομαστική ψηφοφορία. Μπορείτε να ψηφίσετε τώρα. Τελική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες και εγκρίθηκε 37 ψήφι περ 19 κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Κύριε Γιούρεκ, έχετε διαδικαστικό, ε? παρακαλώ, σας ακούμε. έχω την άποψη της ε, μειοψηφίας. Αυτό θέλω να πω για αυτό το ψήφισμα. Πρόεδρος. Βάσει του άρθρου 52 υπάρχει. Και αν είναι κάτω από 100 λέξεις, η γραμματεία θα φροντίσει. Ωραία, έχουμε και άλλες ψηφοφορίες βέβαια, έτσι δεν τελειώσαμε. Επόμενο σημείο για να ψηφίσουμε είναι για της ΛΥΜΠΕ και πρόκειται για τη συμφωνία των πολιτικών ομάδων για ένα σχέδιο κειμένου για να ολοκληρωθεί η συζήτηση μετά από προφορική ερώτηση για το θέμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τις χώρες μέλη όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια. Μία ψηφοφορία ψηφίζουμε. Ξανά με τις κάρτες σας, έτσι ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Ψηφίζετε όλοι. Εντάξει, μπορεί εγώ να σας έδωσα την τύπωση ότι τελειώνουν οι ψηφοφορίες, αλλά δεν τελειώνουν. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Ψηφίσατε όλοι τώρα. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε 38 υπέρ 16 κατά 2 αποχές. Και εδώ ολοκληρώθηκαν οι ψηφοφορίες. Σας ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι. Συνάδελφοι, το 5 θα το πιάσουμε σε δύο λεπτά, αλλά παρακαλώ, ε, εάν δεν θα μείνετε για αυτό το θέμα, να φύγετε ησύχω. Ευχαριστώ. συνάδελφοι, να καλωσορίσουμε εδώ τον επόπτη για, για την προστασία των ευρωπαϊκών δεδομένων. Ο κύριος Μπουταρέλη θα παρουσιάσει την έκθεση για την ε, online, τη διαδικτυακή υπεξαίρεση και χρήση των προσωπικών δεδομένων Θέλω να τον ευχαριστήσω και, και όλοι μας τη δουλειά κατά την περίοδο πριν αρχίσει να ισχύει το GDPR που έγινε πραγματικότητα πριν λίγες εβδομάδες. Χωρίς καθυστερήσεις, Τζοβάνι θα σου δώσω το λόγο για μια δεκάλεπτη παρουσίαση. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, περιτώ να πω ότι είναι μεγάλη μου χαρά να σας μιλώ σήμερα το απόγευμα. Δεν είναι σύμπτωση που το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη έχει προγραμματιστεί λίγο πριν την ακρόαση που διοργανώνει με την ΑΦΚΟ και την Γιούρη η Επιτροπή σας. Στην ε, εργαζόμαστε επί της ομοδότησής μας για την διαδικτυακή υπεξαίρεση προσωπικών δεδομένων προτού η περίπτωση Facebook και Cambridge Analytica βγει στα πρωτοσέλιδα. Μετά το Mini G7 στη Ρώμη και μετά την Ταορμίνα πέρσι συνειδητοποιήσαμε ότι το θέμα των ψευδών ειδήσεων είχε να κάνει και με διαρκή χρήση, ε, παράνομη χρήση προσωπικών δεδομένων πολλών πολιτών συστηματικά. Υπό το φως ε, του σκανδάλου δεν χρειάστηκε βέβαια επικαιροποίηση, διότι το πρόβλημα της ε, διαδικτυακής παράνομης χρήσης δεν έχει απλώς να κάνει με πρακτικές κάποιων ιδιωτικών εταιριών, έχει να κάνει με πρακτικές που είναι κατά πάσα πιθανότητα παράνομες και σίγουρα αντιδιοντολογικές. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο τα κοινωνικά δίκτυα και το περιεχόμενό τους. Δεν είναι αυτή η ιστορία. Δεν πρέπει το θέμα να το κάνουμε κάτι τόσο τετριμένο και να το αντιμετωπίσουμε έτσι. Έχουμε να κάνουμε με όλο το οικοσύστημα των ψηφιακών πληροφοριών το οποίο ε, ήταν ελεύθερο και μεγάλωσε χωρίς νομικούς περιορισμούς. Ε, εξαπλώθηκε κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι λοιπόν στρατηγικό το ζήτημα για τι αρχέ προστασία προσωπικών δεδομένων ήδη από την εφαρμογή τη ισχύω του GDPR. Ε, και αυτή η γνωμοδότηση ήταν προτεραιότητα για μένα παρά την έλλειψη πόρων που υπάρχουν στην αρχή μα. Λίγα δεδομένα λοιπόν για την κατάσταση όπω έχει διαμορφωθεί σήμερα. Πρώτον, το συμπέρασμα ότι ένας μικρός αριθμός ε, γιγαντιαίων εταιριών έχουν ε, αναδυθεί ω κάτοχοι ψηφιακού περιεχομένου που καταναλώνει ο κόσμο είναι σαφέ. Έπειτα, τρία τέταρτα των Ευρωπαίων χρησιμοποιούν το διαδίκτυο παρά την τηλεόραση ή τι εφημερίδε για την άντληση πληροφοριών. Τρίτον, οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή κάνουν αναζητήσεις στο διαδίκτυο μέσω των εφιών τηλεφώνων, όπου το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς το έχουν αυτές οι γιγαντιαίες εταιρείε και μετά οι περισσότερες διαφημίσεις πηγαίνουν στις μεγάλες πλατφόρμες παρά στην τηλεόραση. Άρα ε, φτάνουμε σε δαπάνες ύψους του ΑΕΠ στους κάτους μέλους, της Μεγάλης Βρετανίας. Ε, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτό το γεωπόλιο, όπως έχει ονομαστεί οι διαφημιστές. Και δεν ξέρουμε για τι κάποιε συγκεκριμένε θέσεις στην οθόνη των πλατφορμών αποδίδονται σε συγκεκριμένε διαφημίσεις. Πάντως, το που εμφανίζεται το περιεχόμενο καθορίζεται από αλγόριθμους Πότε το περιεχόμενο που μπορεί να είναι ρατσιστικό πόλωσης ε, ή εκφράζει θυμό μπορεί να προβάλλεται μόνο και μόνο γιατί φέρνει εισόδημα. Οι επενδύσεις στις νεοφύης επιχειρήσεις μειώνονται διότι οι επενδυτές δεν πιστεύουν στον ανταγωνισμό σε σχέση με τις εταιρείες που δεσπόζουν στην αγορά και το σύστημα αυτό έχει προκαλέσει το μεγαλύτερο πρόβλημα στην προστασία των δεδομένων, την ιδιωτικό βίο και την προστασία της ελευθερίας του λόγου έχουμε ανεχθεί πρακτικές εκτός ελέγχου τώρα, διότι όλοι πιστεύαμε ότι είχαν να κάνουν μόνο με τον κόσμο του εμπορίου και των επιχειρήσεων. όμως τελικά χάνουμε τον έλεγχο των δεδομένων μας. Το ίδιο οικοσύστημα έχει αρχίσει να πλήττει τη δημοκρατία και την κοινωνική συνοχή. Προσέξαμε ότι η ανθρωπινά αυστηρή σε τρία επίπεδα μάλλον είναι θύματα σε τρία επίπεδα. Πρώτα απ' όλα παρακολουθούνται όποτε συνδέονται. Δεύτερον, κατηγοριοποιούνται με τρόπους που εμείς δεν μπορούμε να τους αντιληφθούμε και να τους αμφισβητήσουμε και έπειτα τους ε, παρέχονται πληροφορίες βάσει αλγορίθμων ανάλογα με το τι παράγει το μεγαλύτερο κέρδος. Αυτό δίνει μια ψευδέστηση ελευθερίας του λόγου και το να επικεντρώνουμε την δύναμη της πληροφόρησης σε λίγα χέρια όπως αυτή η πρακτική ε, δίνει το δικαίωμα σε δόλιους ε, ε, δρόντες να πάρουν τον έλεγχο της κατάστασης όπως το δημόσιο χώρο. Αυτό που έμοιαζε με χώρους, με φόρα ελεύθερης έκφρασης τελικά γίνονται τόποι και χώροι όπου οι πληροφορίες διαστρεβλώνονται. Είναι αντικείμενο διαστρέβλωσης. Έχετε ακούσει πώς μπορεί κανείς να παίξει με τους αλγοριθμούς για να, να ε, προλάβει ένα κακό αποτέλεσμα. Οι αλγόριθμοι μπορούν να ε, προγραμματιστούν και να προκαλέσουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Άρα πρέπει να μας απασχολήσει τι είναι το διοντολογικό. Τι είναι αυτό που θα πλήξει λιγότερο τους άλλους, είτε είναι καταναλωτές, εργαζόμενοι ή κάτι άλλο. Η δεοντολογία θα έπρεπε να προβλέπει ότι και να θεωρεί μια συγκεκριμένη συμπεριφορά λανθασμένη, ακόμη και αν υπάρχει κατ' επίφαση ε, συμμόρφωση με τον νόμο, όπως στην περίπτωση του GDPR. Τώρα με το GDPR και το EDPP οι επιχειρήσεις πρέπει να αρχίσουν να ενστερνίζονται το πνεύμα του νόμου, δηλαδή να προστατεύουν τους ανθρώπους, όχι τους ε, ελεγκτές, όπως ε, θα συμπεραίναμε με τα σημειώματα που έχουμε λάβει όλοι τις τελευταίες μέρες. Και ταυτόχρονα μπορούμε και εμείς να αναθεωρήσουμε αυτή τη στιγμή την άδικη ε, κατανομή του ψηφιακού μερίσματος τα κοινοβούλια που λογοδοτούν στους πολίτες, όπως το κοινοβούλιο σας, θα πρέπει να αποστείλουν ένα μήνυμα προς τις εταιρείε ότι τελικώς δεν είναι υπόλογες μόνο στους μετόχους τους. Ε, γι' αυτό δεν πρέπει να γοητευτούμε από τις ε, κατ' επίφαση δικαιολογίε των ε, θέμετων πρακτικών και όσων τις ε, θέτουν σε εφαρμογή θα πρέπει το τι είναι διντολογία και τι θα πρέπει να ισχύει με το GDPR και όλες αυτούς τους κανόνες να κανονίζεται από το νόμο με δημοκρατικές διαδικασίες, όχι από τις κερδοσκοπικές εταιρείε. Ε, με όλα αυτά παραμένω στη διάθεσή σας για περισσότερη συζήτηση και διάλογο και με την αρχή μας θα προσπαθήσουμε να υποστηρίζουμε τις υπηρεσίες ε, πληροφοριών και προστασίας δεδομένων της, ε, του ΕΒ Βασιλείου και άλλων διότι η έρευνα αυτή είναι ζωτική σημασία. Το ζήτημα αυτό άλλωστε θα συζητηθεί και στην επόμενη ολομέλεια του EDPP στις αρχές Ιουλίου, όπως θα σας πει και ο συνάδελφός μου, Αντρέη, εντό ολίγου, και δεν μπορώ παρά να τονίσω ότι το μήνυμά μου σήμερα είναι κρίσιμο αλλά ό,τι και να αποφασίσετε υπό το φως της υπόθεσης ε, Facebook Cambridge Analytica θα επηρεάσει το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα χειριστεί τις μεγάλες υποθέσεις και προκλήσεις που θα προκύψουν τα ερχόμενα 5 και 10 χρόνια. Πλησιάζουν οι ευρωεκλογέ. Νομίζω ότι αυτήν την χρονική συγκυρία πρέπει να την προσεγγίσουμε προβάλλοντας τις σωστές ε, προβλέποντας μάλλον τις σωστές εγγύησεις ώστε να προστατευτούν όλα τα πολιτικά κόμματα και όλες οι φωνές. Γι' αυτό πρότεινα στους συναδέλφους μου στην EDPD ε, μετά τον πρώτο γύρο συμπερασμάτων από την υπόθεση Facebook Cambridge Analytica να δούμε κατά πόσον μπορούμε να προτείνουμε κατευθυντήριε γραμμές για τις πολιτικές διαφημίσεις και τις προεκλογικές εκστρατείες. Θα πρέπει αυτό να είναι μια προτεραιότητά μας ε, μέχρι το τέλος του 2018. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε Τζοβάνι. Βεβαίω και γι' αυτό σου ζητήσαμε να μιλήσει πριν την ακρόαση για την Facebook Cambridge Analytica και τώρα έχουμε λίγο χρόνο για ερωταπαντήσει. Η Μπάρμπαρα Σπινέλη πρώτη. Ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον δόκτορα Μπουταρέλη για τη γνωμοδότηση αυτή. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Έχω μια ερώτηση για την συνεργασία που αποτελεί και αντικείμενο σύσταση στην γνωμοδότηση για το πώς η ραδιοτηλεοπτικοί φορείς και οι εκλογικοί παρατηρητές μπορούν να συνεργαστούν. Τι ακριβώς εννοείται λοιπόν με αυτή τη μορφή συνεργασίας. Δεν υπάρχει κίνδυνος μιας removal, κατάργησης περιεχομένου, ψηφιακού περιεχομένου που δεν ε, είναι έγκυρεο. Μπορούμε να βάλουμε στο ίδιο, να δώσουμε την ίδια αξία στις διαφημίσεις και στην γνώμη του πολίτη που ψηφίζει και επίσης για τη δυνατότητα αντίδραση όταν παραβιάζεται ο δυτικό βίος. Το GDPR τώρα το επιτρέπει, όμως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει διαφορετική άποψη για τον ορισμό που ζητούσαν οι καταναλωτέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ζήπελ. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον κύριο Γκουταρέλη για την ε, ανάπτυξη του θέματος. Νομίζω ότι όλες και όλοι έχουμε αντιληφθεί ότι δεν πρόκειται μόνο για την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων, αλλά κυρίως η δυνατότητα δημιουργίας προφίλ στην βάση των δεδομένων αυτών που είναι το πρόβλημα, διότι με τη δημιουργία των προφίλ πράγματι μπορεί να προκύψει και οικονομικό όφελος σε ό,τι αφορά τη στοχευμένη διαφήμιση, αλλά και κοινωνικοπολιτική επιρροή με τρόπο που ο φυγόμενος δεν μπορεί καν να αντιληφθεί ότι επηρεάζεται, διότι αυτοί που στην ουσία τον κατευθύνουν, τον χειραγωγούν, δεν εμφανίζονται ως εκπρόσωποι κάποιου συγκεκριμένου πολιτικού σχηματισμού. Είναι λοιπόν σωστό να επισημάνουμε και πάλι ότι ο βασικός κανονισμός προστασίας δεδομένων δεν αποτελεί μόνο διεθνές πρότυπο προστασίας δεδομένων, αλλά πρέπει να εφαρμοστεί κυρίως και ιδίω να εφαρμοστεί συνεπώ και θεωρώ ότι εν προκειμένου πρέπει να παίξει ρόλο η δέσμευση για την χρήση των δεδομένων καθώς και η ενίσχυση των αρχών προστασίας δεδομένων ώστε να μπορούν να παίξουν σωστά τον ελεγκτικό ρόλο τους. Σε ό,τι αφορά την χειραγώγηση, είτε πρόκειται για οικονομικούς είτε πρόκειται για πολιτικούς σκοπούς, εκεί μπαίνουμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο έχει μεγάλη σημασία, δηλαδή αυτό που λέγεται στα αγγλικά e-privacy. Οι επικοινωνίες δηλαδή μεταξύ δύο μερών πρέπει να προστατεύονται ανεξαρτήτως περιεχομένου. Δυστυχώς, εξ όσων γνωρίζουμε μέσα από την τρέχουσα συζήτηση, είναι μια υπόθεση την οποία τροχοπεδεί, φρενάρει το Συμβούλιο. Δεν έχει αντιληφθεί την βασική σημασία για την δημοκρατία. Θέλω να κάνω μία παρατήρηση ακόμη. Χαίρομαι που στην ακρόαση για το Facebook συμμετέχουν και συνάδελφοί μας από άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές, διότι το πρόβλημα το οποίο θέτει ο κ. Μπουταρέλη δεν αφορά μόνο τα λεγόμενα κοινωνικά δίκτυα, αναφέρεται σε όλους τους stakeholder που συλλέγουν πλήθος δεδομένων Facebook, Google, Amazon, και κατά βάση θεωρώ πρόκειται για ένα πρόβλημα Εάν δηλαδή είναι πάντοτε σωστό να θεωρεί κανείς ότι οι τέτοιες επιχειρήσεις πρέπει να επιτρέπεται να γίνονται όλο και μεγαλύτερες, να καταλαμβάνουν μονοπωλιακές θέσεις, να αποκλείεται εν τέλει ο ανταγωνισμός, πρόκειται για, μια, για ένα θεμελιώδες πρόβλημα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Τελευταία παρατήρηση. Εάν πρόκειται να θεσπίσουμε νέους κανόνες, θα πρέπει σε αυτούς να περιληφθεί και κάτι που συζητείται τώρα πολύ. Δηλαδή, μέσω του φορολογικού δικαίου, πέραν της προσθέσεως των δεδομένων, πρέπει να περάσει και από μία μεταρρύθμιση του φορολογικού δικαίου. Πρέπει δηλαδή να σκεφτούμε και άλλους τρόπους διασφάλισης θέμη του ανταγωνισμού και στο ψηφιακό πεδίο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Μπρικίτε. Εσείς. Όλμπρεχτ. Είναι η τελευταία συνάντηση της Επιτροπής Λίμπε στην οποία συμμετέχω. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κύριο Μπουταρέλη και την ομάδα του που συνεργάστηκαν τόσο στενά μαζί μας για τα θέματα αυτά. Και βεβαίως ευχαριστώ και όλους και όλους τους συναδέλφους με τους οποίους έχω συνεργαστεί εδώ θα ήθελα ωστόσο να προσθέσω ακόμη μία ερώτηση όσον αφορά το θέμα που ήδη αναφέρθηκε σχετικά δηλαδή με τους πόρους των εποπτικών αρχών. Το ερώτημα εάν υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας όχι μόνο μεταξύ αρχών προστασίας δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά σε ό,τι αφορά την εποπτεία και επιβολή του νόμου διεξαγωγή ερευνών στενότερη συνεργασία με αρχές προστασίας δεδομένων και ασφάλειας ηλεκτρονικών δικτύων και ενδεχομένως και με αρχές εποπτείας των μέσων στις χώρες μέλη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Γιάν. Σου σε έχουμε ήδη αποχαιρετήσει με στο Twitter και email κλπ. Δεν τα είπαμε βέβαια και προσωπικά χωρίς να θέλω να σε κάνω να θεωρώ ότι θα είσαι μεγάλη απώλεια για την Επιτροπή Θεμελιωδών Ελευθεριών. Έχει συμβάλει πολύ σημαντικά και απευθυνόμενος προσωπικό, προσωπικός σε σένα, ξαναλέω ότι η αποχώρησή σου είναι μεγάλη απώλεια, διότι η παρεμβάση σου ήταν πάντοτε εξαιρετικής ποιότητας. Ευχαριστώ για την εργασία που έχει καταβάλει στην παρούσα Επιτροπή. I really hope you're going... Σου έχω πει τρεις φορές ευχαριστώ στο Twitter έως τώρα. Ελπίζω ότι θα μπορέσει να φύγει σήμερα. Για να μην συνεχίσω, ε, το εννοώ βεβαίω ε, πάρα πολύ ευγενώ. Θα σε ε, νοσταλγήσουμε, είμαι σίγουρο. Η κυρία Άννα θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Μπουταρέλη και την ομάδα EDPS για τη σημαντική τους συμβολή. Όταν ξέσπασε το σκάνδαλο Cambridge Analytica, ήρθε ο κ. Μπεταρέλη εδώ και μας είπε πρόκειται για το σκάνδαλο του αιώνα. Και σήμερα πράγματι μας εξήγησε με περισσότερες λεπτομέρειες γιατί το είπε αυτό. Πρόκειται για σημαντική πρόκληση για μας τους εκλεγμένους εκπροσώπους και νομοθέτες, αλλά από την άλλη μεριά γνωρίζουμε και τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουμε. Ρωτώ, συμφωνεί ότι ένα κρίσιμο στοιχείο για να μπορέσει να ε, σπάσει αυτή η κυρίαρχη θέση είναι μέσω της φορολογίας. Κάτι που πρέπει, οφείλουμε να απαιτήσουμε από τις κυβερνήσεις των χωρών μας να λάβουν αυστηρότατα φορολογικά μέτρα εις βάρος αυτών των ψηφιακών πλατφορμών. Εποφελία των κρατών και βέβαια των πολιτών τους. Ρωτώ, είπατε ότι οι αλγόριθμοι μπορούν να προκαλέσουν διοντολογικές ανησυχίε. Τι γίνεται όμως με την τεχνητή νοημοσύνη. Διότι βεβαίως εκεί η δυνατότητα να ενταχθεί ας πούμε μέσα στην ε, τεχνητή νοημοσύνη η, μια διάσταση ε, διοντολογίας ε, πρόκειται στην ουσία για οξύμορον. Θα, δεν θα είχε πολύ καμία διάσταση διοντολογική. Διάβασα σήμερα ότι το Facebook ήδη χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να επισκευάζει εντό εισαγωγικών κάποια προβλήματα εμπορικού χαρακτήρα. Τώρα, άλλο θέμα, δεν ξέρω αν ο κ. Μπουταρέλη θα ήθελε να μας πει κάτι σχετικά. Είδαμε ότι αυτή η υπόθεση Cambridge Analytica είναι η κορυφή του παγόβουνου. Γνωρίζουμε τώρα ότι αυτή η Cambridge Analytica διασυνδέεται με άλλες επιχειρήσεις. Αυτές δηλαδή που επενδύουν στην χειραγώγηση εκλογών με ευνοϊκό αντίκτυπο βέβαια μετά και στις επιχειρήσεις αυτές. Όπως η επιχείρηση ένι και, ε, και εταίροι, ένι και partners, που δεν δραστηριοποιούνται μόνο στη Μάλτα, αλλά και αλλού. Και είδαμε ότι έχουν, συνδέονται με την Cambridge Analytica. Και βέβαια και οι δικηγορικές εταιρείες οι οποίες εμπλέκονται με τέτοιες επιχειρήσεις που διώκουν δημοσιογράφους οι οποίοι αποκαλύπτουν τα δεινά που πράττουν όλοι αυτοί. Και, και ε, δικηγορικές εταιρείε οι οποίες έχουν την έδρα τους στη Βρετανία, όχι μόνο, που προβαίνουν σε δράσεις SLAP, δηλαδή ε, προληπτικές αγωγές έτσι ώστε να αποτραπεί η ενημέρωση του κοινού. Μήπως να αφήσετε λίγο καιρό στον Ζωβάνι να μπορέσει να απαντήσει, λέει ο πρόεδρος. Και εγώ τον ερωτώ. Γνωρίζετε τι γίνεται, πώς αντιδρούν οι εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων σε αυτά τα μεγάλα θέματα και είναι και το θέμα βέβαια στην ε, Μεγάλη Βρετανία. Νομίζω ότι εκεί η αρμόδια αρχή αντιδρά σωστά. Αλλά έχετε κάποια γενικότερη άποψη σχετικά με το πώς αντιδρούν οι εποπτικές αρχές σε όλη την Ένωση και Ιδίω στη βάση του EDPS καθώς τα θέματα αυτά γίνονται πιο έντονα και πολιτικά πιο δύσκολα. μπορείτε να απαντήσετε. Um, Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω και θα ξεκινήσω από την κυρία Σπινέλη. Όταν πριν από ένα χρόνο ξεκινήσαμε την πρωτοβουλία μας για το Digital Clearing House, είχαμε διάφορες συναντήσεις με αρμόδιους και υπεύθυνους όσον αφορά την προστασία των δεδομένων και ξέραμε ότι όλοι είχαν να παίξουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο και καταλάβαιναν ότι θα έπρεπε να μην υπάρχουν επικαλύψεις Υπάρχουν οι αρμόδιοι εθνικό επίπεδο για αντιτράστ που ασχολούνται κυρίως με το θέμα της ε, βασικής συλλογής προσωπικών δεδομένων. Εμείς θέλουμε λοιπόν να συγχρονίσουμε τους φακέλους μας και η επόμενη συνάντηση του φόρουμ αυτού θα συμπεριλάβει και τους ρυθμιστές όπου σε μερικές χώρες είναι και οι αρμόδιοι προκειμένου να τηρήσουν την αρχή των ίσων ευκαιριών. Ακριβώς επειδή ασχολούνται με τα οπτικοακουστικά. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι αυτό θα οδηγήσει σε κάποιο είδους λογοκρισία. Τώρα, κατά τα άλλα, ο κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ε, περιλαμβάνει διάφορες έννοιες αλλά και κάποιους προορισμούς παρά το γεγονός ότι προσπαθήσαμε να πάμε όσο γίνεται πιο μακριά. Καλύφθηκαν πολλά κενά, αλλά σίγουρα όχι όλα στον τομέα της προστασίας των δεδομένων. Πάντως, οι διατάξεις όσον αφορά την βλάβη ή την ε, δικαστική διόρθωση, αποζημίωση. Ευχαριστώ την κυρία Σίπελ για την ερώτηση που έκανε όσον αφορά την ιδιωτικότητα, γιατί αυτό μου επιτρέπει να πω μην αναβάλλεται για το 2020 αυτό το φάκελο. Όπως ε, λέμε στον κανονισμό μας, το θέμα της προστασίας του ιδιωτικού βίου δεν είναι απόλυτα καλυμμένο. Και σίγουρα υπάρχει θέμα θεμητού συμφέροντος και ανάλογα με αυτό προβλέπονται οι διατάξεις για τις επιχειρήσεις. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε να παραμένουν κενά και να μην είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα των πολιτών για άλλο λόγο πέρα από αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεχθεί οι εταιρείε, οι επιχειρήσεις ή οτιδήποτε ε, που γνωρίζει ο πολίτης ότι έχουν τα δεδομένα του. Πρέπει λοιπόν ο κόσμος να είναι σε θέση να έχει καλύτερα τα δεδομένα του και να υπάρχουν κίνητρα για την αγορά να καινοτομήσει. Όχι βάσει των παλιών ε, προτύπων, αλλά να έχουν στη διάθεσή τους εργαλεία ώστε όλοι οι άνθρωποι να μπορούν να ελέγχουν τη ζωή τους και τα δεδομένα τους. Δεν μπορούμε στην Ευρώπη να ισχυριζόμαστε δράσεις όσον αφορά την περίπτωση της Cambridge Analytica εφόσον δεν έχουμε εμεί τη σωστή εικόνα, δεν την έχουμε φτιάξει για την προστασία των δεδομένων. Τώρα Γιάννη ευχαριστώ για την ερώτηση. Όντω, πολλές φορές έχουμε πει πόσο καλό ρόλο έχει παίξει όλα αυτά. Οι αρμόδιες αρχές συντονίζουν πάρα πολύ. Και το νομικό σύστημα πολλών χωρών μελών προβλέπει ήδη την πλήρη χρήση και την υποχρεωτική συνεργασία με άλλες αρμόδιες αρχές. Οι εθνικές διατάξεις προβλέπουν τη δυνατότητα οι επόπτες δεδομένων να συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές. Αυτό που εγώ βλέπω να λείπει είναι πόροι για νέες τεχνολογίες. Οι επόπτες δεδομένων θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιήσουν νέες τεχνολογίες, να είναι φοδιασμένοι δηλαδή, για να μπορούν να κάνουν έρευνες με πιο περίπλοκα εργαλεία. Μίλησα με την Έλισσα Μπεθέγκνη που στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη συνάδελφό μου, και είδαμε ότι από την ανάλυση χιλιάδων φακέλων φαίνεται ότι χρειάζονται και επαρκή σπόροι αλλά και ικανότητες. Και αυτό είναι που αποτελεί πρόκληση για το μέλλον. χρειαζόμαστε παραπάνω 25% πόρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους αρμόδιους επόπτες δεδομένων. Πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο λοιπόν στις νέες τεχνολογίες, στον έλεγχο των εξελίξεων. Χρειαζόμαστε επιστήμονες που να είναι εκπαιδευμένοι στο θέμα των δεδομένων. Κύριε Γκόμες, ευχαρίστω να σας απαντήσω για τη φορολόγηση, αλλά κάποιο θα μου πει «Εσένα η δικιά σου είναι η προστασία των δεδομένων και όχι φορολογία». Θα μπορούσε να βοηθήσει ίσως, ναι, αλλά ειλικρινά δεν είμαι εμπειρογνώμων. Και βλέπω ότι υπάρχει μια κατακαιρματισμένη προσέγγιση από πλευρά των χωρών μελών. Και αυτό είναι πρόβλημα. Προσωπική μου όμως άποψη είναι ότι έτσι όπως προχωράμε είναι σε βάρος των πολιτών και τελικά αφήνουμε έτσι οι έσοδα να φορολογούνται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τους αλγόριθμους, επιτρέψτε μου να πω ότι ναι, υπάρχει περιθώριο. θα έχουμε τον Οκτώβριο που μας έρχεται τους επόμενους Ολυμπιακούς δεδομένων με εκπροσώπους από 81 χώρες. Και φέτος η συζήτηση θα είναι όσον αφορά την ψηφιακή ηθική. Οι αρχές προστασίας δεδομένων, εμείς δηλαδή πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά, πρέπει να ακολουθήσουμε ένα σωστό business model και να δούμε τι βήματα θέλουμε να κάνουμε πλησιάζοντας την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, όπου χρειάζεται περισσότερη αξιοπρέπεια και μεγαλύτερο περιθώριο για τους πολίτες και τους πελάτες. Να δούμε τι ηθικά στέκει και τι όχι, και όχι μόνο νομικά τη στέκει. Πρέπει επίσης βάσει αυτής της εμπειρίας που θα έχουμε περί ηθικής, να δούμε ποιες είναι οι αρχές εκείνες που θα έπρεπε να τηρούνται και ποιος είναι αρμόδιος γιατί. Συγχρόνως η αρχή της προστασίας του ιδιωτικού βίου που προβλέπεται στον ε, νέο κανονισμό για την προστασία δεδομένων σίγουρα θα βοηθήσει πολύ. θα δοθούν κάποια έντυπα με ερωτήσει σε διάφορες αρμόδιες αρχές και προσπαθούμε να πείσουμε όλες τις αρμόδιες αρχές απανταχού να ασχοληθούν περισσότερο με το θέμα αυτό της σχέσης της ηθικής με την ε, τεχνητή νοημοσύνη. Ευχαριστώ όταν έχουμε τα αποτελέσματα να σας τα παρουσιάσουμε. Και τώρα πρέπει να έρθω στην τελευταία σας ερώτηση, κύριε Πρόεδρε οι επόπτες προσωπικών δεδομένων θέλουν να μιλούν με μία φωνή. Και ακόμα και πριν από την πλήρη εφαρμογή του κανονισμού για την προστασία δεδομένων είχαμε αρχίσει να ε, συντονιζόμαστε μεταξύ μας και να εντοπίζουμε που συμφωνούμε. Γίνονται και έρευνες εμπιστευτικά και με το Ηνωμένο Βασίλειο συνεργαζόμαστε. σε θέματα έγκαιρης προειδοποίησης προκειμένου να είμαστε έτοιμοι για τα επόμενα βήματα. Η νομική ανάλυση γίνεται όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων, των προηγούμενων οδηγιών για την προστασία των δεδομένων. Τώρα βέβαια θα πρέπει να δούμε ποιες είναι και οι συνέπειες μακροπρόθεσμα του νέου κανονισμού για την προστασία δεδομένων. Ε, νομίζω ότι είμαστε στο σωστό δρόμο και θέλω να σας καθισχάσω και να σας διαβεβαιώσω ότι σε μερικές εβδομάδες θα ακούσετε κάποια προκαταρτικά αποτελέσματα τα οποία θα έρθουν με συνοχή από όλους τους επόπτες προσωπικών δεδομένων της Ευρώπης συνολικά. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ και εσάς και τους συνεργάτες σας για το έργο σας. Ωραία, συνάδελφοι, τώρα θα διακόψουμε για λίγο. Βλέπω μπαίνουν και συνάδελφοι και από τις άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές και θα αρχίσουμε σε λίγο με την δεύτερη ακρόαση. Σε πολύ λίγο για να υποδεχτούμε όλους τους προσκεκλημένους μας.